αύριο θα γίνει την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, όχι αύριο. Η επόμενη συνεδρία είναι αύριο, 3η 9 Φεβρουαρίου, 9 με 12.30